Dear colleagues, good afternoon. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Ας ε, ξεκινήσουμε. Σημείο 1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης. Να σας ενημερώσω για τις εξής αλλαγές. Τα σημεία 17 και 21 θα τα δούμε μετά το σημείο 11 και τα 12 και 13 μετά από το σημείο 19. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Οπότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Εάν δεν λάβουμε αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά της 7ης Δεκεμβρίου εγκρίνονται και περνάμε στο σημείο 3 έχω εδώ την ευχαρίστηση να καλωσορίσω τον κύριο Βασ τον κύριο Τίμερμανς πρώτο την πρόεδρο της Κομισιόν Αρμόδη, για την βελτίωση της νομοθεσίας τις διοργανικές σχέσεις το κράτος δικαίου και τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων για τον παραδοσιακό ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή μας. Κύριε Αντιπρόεδρε, είστε ο πρώτος με τον οποίο κάνουμε αυτήν την συζήτηση φέτος. Θα συναντηθούμε αύριο με την κυρία Γιούροβα και ελπίζουμε τον Μάιο με άλλους επιτρόπους. Τα χαρτοφυλάκια των οποίων αφορούν τις αρμοδιότητές μας, οπότε προτείνω τώρα να λάβετε τον λόγο να μας πείτε πώς έχετε και μετά περνάμε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Να ξεκινήσω με τα φρέσκα. Η πρωτοβουλία για την προστασία των καταγγελόντων νομίζω ότι πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο το καιρό. Και νομίζω ότι χρειάζονται οι καλύτερη προστασία σε κοινοτικό επίπεδο για να υπερασπιστούμε και την ε, κοινή αγορά και την ελευθερία των ΜΜΕ. Οι άνθρωποι αυτοί δίνουν πληροφορίες, κατά το οποίο οδηγεί σε έρευνα, σύλληψη και δίωξη παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου. Επιπλέον, η προστασία τους βοηθά τον να με την ελευθερία της έκφρασης και τον ΜΜΕ. Οι καταγγέλλοντες είναι μια κρίσιμη πηγή ε, της δημοσιογραφικής έρευνας και έχει μεγάλη σημασία για την δημοκρατία. Είναι πυλώνας της δημοκρατίας τα ελεύθερα μηνύα όπως επίσης και η πρόσβαση στις ε, πληροφορίες και άρα είναι πολύ σημαντικοί οι καταγγέλλοντες σε αυτό το πλαίσιο. Προτείναμε υψηλά ελάχιστα ελάχιστες προδιαγραφές ε, προστασία των καταγγελόντων σε πολλούς κλάδους όπου μπορεί να προξενήσει βλάβη στο δημόσιο συμφέρον η παραβίαση του κοινωτικού δικαίου και βεβαίως ε, η προστασία των καταγγελόντων είναι απαραίτητη για να υπάρξει εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα προστατεύσει και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και θα συνεισφέρει σε μια δίκαιη και λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Θα ανοιχνεύσουμε καλύτερα παράνομες ενέργειες, απάτη, φοροδιαφυγή και πρακτικές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον. Έτσι νομίζω σας απαντάμε. Το ζητούσατε εδώ και καιρό, το γνωρίζω. Θεωρώ λοιπόν και έχετε ε, πέρασει και ένα ψήφισμα και στις 19 Απριλίου και νομίζω ότι επιτέλους κάναμε αυτό το οποίο θέλατε. Αυτό ήταν ο στόχος μα. Ότι δηλαδή καταγγέλλοντες ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης θα έχουν διάβλους για να καταγγείλουν εσωτερικά εντός του οργανισμού, εξωτερικά στις αρχές ή δημοσίως μέσω των ΜΜΕ τις πληροφορίε που έχουν. Και τώρα πρέπει ακριβώς να αποφασίσουμε το τι θα γίνει στην περίπτωση που θεωρούν ότι α, ο δικός τους οργανισμός δεν μπορεί να δώσει λύση, προφανώς να έχουν τη δυνατότητα άλλων διάβλων. Οι αρμόδιες αρχές θα είναι υποχρεωμένες να δώσουν συνέχεια στις καταγγελίες αυτές. Η αντεκδίκηση με οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται και τιμωρείται εάν υποστούν αντίπεινα, έχουν ε, διάφορους τρόπους να προσφύγουν ε, ε, παραδείγματος κάνει κατά της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας ή να μην υπάρχει δυνατότητα απόλυσης όσο διαρκεί η διαδικασία στο δικαστήριο. Και εδώ πέρα υπάρχει βεβαίω και το βάρος της αποδείξεως. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δράει βάρος του καταγγέλντος θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν το κάνει για λόγους αντεκδίκησης. Βεβαίως μιλάμε για υπεύθυνε ε, τέτοιες καταγγελίες και στόχο έχουμε να αποθαρρύνουμε την κακόβουλη τέτοια ενέργεια. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να στήσουν επαρκή πλαίσια για την προστασία των καταγγελόντων και να επεκταθούν αυτές οι αρχές και σε άλλους τομείς. Ε, και ζητάμε, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν αυτές τις διατάξεις και στο εθνικό τους δίκαιο. Και βεβαίως αν εγκριθεί η οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί και στο εθνικό πλαίσιο. Τώρα Έχουμε την πρωτοβουλία εταιρικού δικαίου για να βελτιωθούν οι κανόνες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά για να γίνει πιο δίκαιη η κοινή αγορά και να ταιριάζουν οι κανόνες του εταιρικού δικαίου στον ψηφιακό κόσμο. Ελπίζω να εγκριθεί λοιπόν αυτό το Σώμα των Επιτρόπων τις επόμενες ημέρες. Περιέχει δύο προτάσεις, μία αφορά για την ψηφιοποίηση του εταιρικού δικαίου και μία για τις δύο συνοριακές δραστηριότητες. Με την πρόταση αυτή σκοπεύουμε οι επιχειρηματίες ε, να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές στο διαδίκτυο και τα σχετικά ψηφιακά εργασία, εργαλεία με και βεβαίως ε, να υπάρχει η δυνατότητα να αποφευθεί η κατάχρηση ενώ η συνεργασία των εταιριών θα απαιτηθεί και στον εξυγχρονισμό των κανόνων ε, και στην χάραξη κανόνων για τις δύο συνοριακές συγχωνεύσεις. Αναμένουμε βεβαίως ε, να ληφθεί υπόψη το ότι λάβαμε σοβαρά υπόψη μας τα όσα είπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να έχουν μία έδρα στην κοινή αγορά και βεβαίω ε, δεν θέλουμε να εμποδίσουμε κάποια χώρα να μεταφέρει την έδρα της αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει κάποια κατάχρηση του φαινομένου, δηλαδή όταν κάτι τέτοιο γίνεται για στόχους αποφυγής ή αποφυγής των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τέλος ή αποφυγής των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τα λοιπά. Βεβαίως η εσωτερική αγορά μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς μόνο εάν υπάρχει η απαραίτητη εμπιστοσύνη ότι δεν θα υπάρξει κατάχρηση των ευκαιριών που προσφέρει στις επιχειρήσεις. Δεν θέλω να μακρηγορήσω τώρα. Έχω πολλές σημειώσεις εδώ αλλά έτσι δεν θα μπορέσετε να μου κάνετε ερωτήσεις. Μου έχουν πει λοιπόν διάφορα εδώ πέρα για την πρωτοβουλία κράτους δικαίου, για την καλύτερη νομοθεσία, για αναλογικότητα, επικουρικότητα. Μπορώ να τα πω όλα αυτά, αλλά καλύτερο είναι να μου κάνετε εσείς ερωτήσεις και θα επανέλθω σε αυτά με βάση τις ερωτήσεις σας, γιατί οπωσδήποτε θα σας ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα. Συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ναι, ναι, αργήσαμε να ξεκινήσουμε, οπότε είπα να μην μιλήσω άλλο να σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις. Όταν πείτε επανέλθετε στο τάδε ζήτημα, θα το κάνω ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χαουτάλα πρώτα, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Αντιπρόεδρε. Εδώ είμαι. Ναι, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Πρώτον, η Επιτροπή μας και ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένω μέχρι τώρα έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει έναν κανονισμό, μια ρύθμιση για μια ανοιχτή διοίκηση με διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι καλές πρακτικές διοικητικές πρέπει να κωδικοποιηθούν στην ενωσιακή νομοθεσία. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εκείνη είναι που μπορεί έτσι να εγγυθεί τις επιχειρήσεις, ε, τις δουλειές του κόσμου με έναν αποτελεσματικό και ανοιχτό τρόπο. Όμως είναι απογοητευτικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι δεν συμφωνεί με τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχουν αυτέ οι εγγυήσει. Ήδη τον Οκτώβριο του 2016 είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχει πιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται ένα νομοθετικό μέσο. Τώρα, με ιδιαίτερη χαρά, μπορώ να σας πω ότι είμαστε καθοδόν να σας πείσουμε. Γιατί είχαμε μια διαβούλευση με το κοινό ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα ολοκληρώνεται η έκθεση αντικτύπου, όπου συμπεριλαμβάνονται όλε οι αρχέ που υπογραμμίσατε κι εσεί. Θα δημοσιοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα και θα έχουμε εδώ στην Επιτροπή αυτή νομικών υποθέσεων το καλοκαίρι μια ακρόαση. Και είναι προνομιό μου να σας προσκαλέσω, να σας ζητήσω να έρθετε εσείς προσωπικά στην ακρόαση αυτή. Αυτό ήταν το ένα μου θέμα. Δεύτερον, όχι, απαντάτε. Το δεύτερο θέμα μου έχει να κάνει με την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου του Καπιτάνη κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ξέρω ότι έχει να κάνει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια που είναι διαμεσολαβήτρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον τριμερή διάλογο. Και ρωτάω λοιπόν, εσείς πώς εκτιμάτε τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής που ζητάει να υπάρχει πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του τριμερούς διαλόγου, του εκάστοτε τριμερούς διαλόγου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει έφεση, ελπίζω όχι, γιατί νομίζω ότι δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να στείλει στο κοινό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δηλαδή δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στη συνέχεια, αν υπάρξει έφεση δηλαδή όχι, νομίζω ότι πρέπει να υλοποιήσουμε αυτή την απόφαση. Οπότε ρωτάω, εσεί και οι υπηρεσίε σα, το όνομα τη καλύτερη νομοθέτηση έχετε σκεφτεί καθόλου πώ θα θέσετε σε εφαρμογή, πώ θα υλοποιήσετε αυτή την απόφαση. Σαραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την πρότασή σας που δημοσιεύτηκε σήμερα για τους καταγγέλλοντες, του whistleblowers είναι κάτι που όντω, επιμόνως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από τότε που υπήρξε η οδηγία για τις απόρριτες εμπορικές συμφωνίες που όντω απειλούν τους ε, καταγγέλλοντες, ε, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ καλό βήμα. Η πρόταση αυτή δηλαδή πάει στη σωστή κατεύθυνση. Όμως θέλω να σας ρωτήσω και κάτι. Είπατε ότι η καταγγέλλονται, αν πιστεύουν ότι οι εσωτερικοί ιδίωδοι στον οργανισμό τους δεν ε, οδηγούν σε αποτελέσματα ή ότι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο μια ανεξάρτητη έρευνα, τότε πρέπει να πάνε σε, εξωτερική, σε εξωτερικές διόδους. Αλλά και εκεί υπάρχουν αρχές και το έχουμε δει με τα LuxLeaks για παράδειγμα, ότι ένας καταγγέλων πρέπει κατευθείαν να μπορεί να πάει στον τύπο, στο κοινό. Οπότε τα εμπόδια που αναφέρονται στην οδηγία είναι πολλά και μεγάλα. Ε, μιλάτε για διαδικασίες που είναι χρονοβόρες, πρώτα τρεις μήνες, μετά επέκταση σε έξι μήνες, μετά πάει σε εξωτερικές διόδους κλπ. Οπότε, και το ξέρετε, πολλές φορές ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο επεκτείνεται συνήθως αποτελεί τον κανόνα και θα έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος προτού να μπορεί ο καταγγέλων να απευθυνθεί στο κοινό και να ζητήσει την κάλυψη από την οδηγία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύουμε τους καταγγέλλοντες όταν πηγαίνουν στο κοινό κατευθείαν και αυτό να μην γίνεται μόνο στην περίπτωση που πρόκειται ελοχεύει κάποιος κίνδυνος για το κοινό. Μόνο τότε. Αλλιώς όλη αυτή η ιδέα της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης καταστρέφεται. Γιατί αν πρέπει να αποδείξει ο καταγγέλλον τον κίνδυνο, ε, δεν βοηθάει. Δεν πρέπει να, πρέπει να το αποδείξουν για να έχουν προστασία. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι θα έπρεπε να βάλουμε σε πιο ισχυρή θέση τον καταγγέλλοντα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, ε, εσείς τι λέτε, ποιος τελικά θα πρέπει να αποδείξει κατά πόσο υπάρχει άμεσος κίνδυνος ή όχι. Και αν πάνε κατευθείαν στο κοινό οι καταγγέλλοντες αντί να πάνε στις αρχές, θα προστατεύονται ή όχι. Ευχαριστούμε κυρία Κάουφμαν. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα φρέσκα που είπατε περί καταγγελόντων και να σας ευχαριστήσω για το ότι κάνατε αυτό το οποίο ζητούσε εδώ και καιρό το Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και ελπίζω τελικά να είμαστε σε θέση και εμείς ως νομοθέτης να εργαστούμε γρήγορα για να τέθει όντως ενισχύ η νομοθεσία αυτή και βλέποντας το κείμενο μπορώ να σας πω ότι πράγματι είναι πολύ φιλόδοξη η πρόταση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις για να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα θέματα του εργατικού δικαίου, παραβιάσεις του εργατικού δικαίου κτλ. Στο μέτρο που μπορώ να κρίνω δεν θα ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής ζητήματα ασφάλειας των τοπαργασίας, υγεία των εργαζομένων. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που ανήκουν σε αυτόν τον τομέα. Και το δεύτερο, εάν κατάλαβα καλά, η πρόταση της Κομισιόν αναφέρεται στο κοινοτικό δίκαιο και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς άνθρωποι οι οποίοι ε, βλέπουν κάτι τέτοιο μπορούν να διακρίνουν μεταξύ εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Γιατί βεβαίως ε, υπάρχουν κάποιες ε, κρίσες ζώνες και θα σκεφτεί βεβαίως ο καθένας ε, πριν δημοσιοποιήσει κάτι τέτοιο πως είναι υπερβολικά περίπλοκο. Κύριος Μπρετό, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σήμερα μας παρουσιάζεται μια πρόταση οδηγίας ενδιαφέρουσα για τους κατακέλοντες είπατε ότι αποτελούν πυλώνα της δημοκρατίας και συμφωνώ με την ανάλυση αυτή. Πράγματι, χρειαζόμαστε ένα αντίβαρο και οι καταγγέλλοντες είναι ακριβώς για να προειδοποιούν κάθε φορά που βλέπουν να υπάρχει κάποια παραβίαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζω ότι είναι σημαντικό και γι' αυτό και ψήφισε την έκθεση Ροζιέ πέρυσι, η οποία ακριβώς ζητούσε τη δικιά σας παρέμβαση. Εγώ ο ίδιο, εκ μέρου τη ομάδα μου στην Ολομέλεια, είχα υποβάλει ένα εναλλακτικό ψήφισμα που πήγαινε όμω προ την ίδια κατεύθυνση προστασία των καταγγελόντων. Δέκα χώρε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχουν μια πλήρη νομοθεσία για να προστατεύουν του ανθρώπου αυτού. Οπότε η δικιά σα παρέμβαση για να οθήσετε τις χώρες μέλη να εμπνευστούν από τα καλά παραδείγματα είναι φυσικά ευπρόσδεκτη. Από την πλευρά μου χαίρομαι που προσπαθούμε να πλαισιώσουμε την διαδικασία καταγγελιών σε τρεις χρόνους από ό,τι κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα για τις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει μια εσωτερική δίωδος, διευθέτηση, η οποία επιτρέπει αν είναι καλή τυπίστη η επιχείρηση να διευθετηθεί το θέμα. Στη συνέχεια προσφυγή σε μια κρατική αρχή και χαίρομαι που περνάμε από τις κρατικές αρχές και σε ένα τρίτο χρόνο, αν αυτό δεν φτάνει, τότε προσφυγή στον τύπο. Οπότε η περίπτωση της άμεσης απειλής και στην περίπτωση που υπάρχει αυτή να μπορεί ο καταγγέλων να προσφύγει στο κοινό κατευθείαν, νομίζω ότι είναι θετικό. Ε, αυτό λέμε και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά και κάτι ακόμα. Βλέπω μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ε, περάσουμε. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε το κείμενο αυτό για να φτιάξουμε μια κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία όσον αφορά την προστασία των καταγγελόντων. Νομίζω ότι θα ήταν μια κακή ιδέα. Αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσουμε πραγματικά όθηση στις χώρες μέλη να αναπτύξουν τη δικιά τους εθνική προστασία. Και το λέω αυτό γιατί στο σημείο 57 της έκθεσης Ροζιέρ υπήρχε αυτή η μνήα. Η δυνατότητα δηλαδή να δημιουργηθεί μια κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία γι' αυτό. Οπότε ρωτάω, είναι στις προθέσεις σας να πάτε προς την κατεύθυνση ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Το θέμα της νομικής βάσης. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το αναφέρατε αυτό καθόλου. Είχαμε μιλήσει επί μακρό στις διάφορες επιτροπές που δούλεψα πάνω στην έκθεση Ροζιέρ. Το σημείο 1 μάλιστα της έκθεσης αυτής υπογράμμιζε ε, με τρόπο όχι ικανοποιητικό, ότι υπήρχαν πολλές νομικές βάσεις χωρίς όμως να λέει ποιες. Οπότε καταλαβαίνετε, για ένα νομικό αυτό φαίνεται πολύ περίεργο. Θα ήθελα λοιπόν εσείς να μας καθησυχάσετε ότι θα καταλήξετε σε μια σαφή νομική βάση για αυτό το κείμενο. Και τρίτον, πιο δυσάρεστο ίσως, η σημερινή σας παρουσίαση με το Σαν Μάρτεν Γκέιτ διότι Επρόκειτο για αυτόν τον ε, Γενικό Γραμματέα που έγινε Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε και γράφτηκε πολύ στον τύπο στις διάφορες χώρες μέλη. Γίνανε πολλές διαμαρτυρίες και εμεί οι ίδιοι γίναμε καταγγέλλοντε κατά κάποιο τρόπο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν οδήγησε αυτό πουθενά. Εσά λοιπόν αυτή η αντίφαση δεν σα ενοχλεί, δηλαδή να μα προτείνετε ένα κείμενο που προστατεύει του καταγγέλλοντε και από την άλλη φορά όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τηρεί τι υποχρεώσει τη, τότε κάνουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Uh, αυτό ήταν ο πρώτο γύρο ερωτήσεων. Οι υπόλοιποι θα υποβάλουν τι ερωτήσει του σε μια επόμενη φάση. Ο κύριος Επιπρόεδρο θα απαντήσει τώρα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσει. Θα απαντήσουμε τη σειρά που υποβλήθηκαν. Για το διοικητικό δίκαιο. Επί μακρόν κάναμε αυτή τη συζήτηση. Η θέση σα δεν άλλαξε, ούτε η δική μου. Μα ξέρετε. Πείστε με αν μπορείτε, αν υπάρχουν νέα επιχειρήματα. Αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έρθω σε μια δική σα ακρόαση και να σα ακούσω, το κάνω ευχαρίστω. Μπορεί και να με πείσετε εσεί ή να σα πείσω εγώ, ποιο ξέρει. Στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, λοιπόν, μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψει. Ο διάλογο δεν γίνεται μεταξύ ανθρώπων που συμφωνούν κατά ανάγκη. Μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Ε, θα δω βέβαια και την ατζέντα μου να δω τι διαθεσιμότητε έχω, αλλά θα κάνω κάθε προσπάθεια για να έρθω. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του δικαστηρίου αυτού και το θέμα των τριμερών διαλόγων, την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του τριαλόγου, αυτό αφορά περισσότερο το Συμβούλιο παρά την Κομισιόν. Θα περιμένουμε τη θέση όμως του Κοινοβουλίου, γιατί δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Δεν ξέρω αν θα κάνει προσφυγή εναντίον της απόφασης στο Κοινοβούλιο. Ε, ελπίζετε όχι, ε? αλλά δεν ξέρετε κιόλα. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να σας πω το εξή. Και εγώ ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι στα πλαίσια του διαθεσμικού διαλόγου που έχουμε για την ε, διαφάνεια. Και ελπίζω αυτό να δώσει καρπούς. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια. Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, αλλά είμαστε φιλόδοξοι εμείς στην Κομισιόν. Αυτά μπορώ να πω από πλευράς Κομισιόν για το θέμα αυτό, προς το παρόν. Ετοιμάζοντας την πρόταση για τους καταγγέλλοντες, πάντα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση για τις διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να δημιουργήσουμε, ούτω ώστε να είναι, μια δίκαιη, να είναι δίκαιη αυτή η προσέγγιση. Πάντα κάποιοι στο κοινοβούλιο λέγανε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία, δηλαδή να γίνει μια μια πρώτη εσωτερική προσφυγή, μετά να πάει το άτομο στους αρχές και τα λοιπά και μετά ε, στον τύπο. όχι, θα πρέπει να μπορεί να πηγαίνει κατευθείαν στον τύπο, να απευθύνεται προς το κοινό, προς τα έξω. Δεν συμφωνώ. Για εταιρείε με παραπάνω από 50 υπαλλήλου. ή τζίρο πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο, πρέπει να δημιουργήσουν αυτή Υπάρχουν οι εταιρείε εσωτερικέ διαδικασίε για του καταγγέλλοντε. Έτσι δημιουργείται μια τελείω νέα δυναμική σε πολλά κράτη-μέλη για εταιρείε που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ίδιε ότι αν υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα θα πρέπει να έχουν διαδικασίε για να το αντιμετωπίζουν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Και μπορεί να αλλάξει τελείω το τοπίο για το πώ λειτουργούν και πώ ε, αποτελεσματικοί είναι οι καταγγέλλοντε. Το ίδιο ισχύει φυσικό, φυσικά και με τι ε, δημόσιε αρχέ. Ε, με τους κρατικούς φορείς. Δεν έχουν όλα τα κρατη διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Δεν τις έχουν ήδη μέχρι να μπει η οδηγία δηλαδή στην εσωτερική νομοθεσία. Τώρα, το τι είναι άμεσος κίνδυνος, ε, αυτό το εκτιμά ο καταγγέλων. Γιατί αν κάποιος έχει το θάρρος να βγει προς τα έξω και να μιλήσει, γιατί θεωρεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται σωστά από την εταιρεία στην οποία εργάζεται ή από τον κρατικό φορέα στον οποίο εργάζεται, ε, τότε αυτή η ηθική επιταγή ε, θα πρέπει να ανταμυφ, ε, που κινητοποιεί τον καταγγέλλοντα, θα πρέπει, να ανταμυφ, θα πρέπει εξαιτία αυτή και χάρη σε αυτή να ανταμυφθεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο καθένα μπορεί να κάνει τι θέλει. Τώρα, η αντιστροφή του βάρου απόδειξη πότε ισχύει. Ισχύει από τη στιγμή που μια εταιρεία τιμωρεί κάποιον επειδή είναι καταγγέλων. Λαμβάνει κυρώσει εναντίον του. Δεν σημαίνει ότι κάποιο ισχυρίζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στην εταιρεία. Τότε η εταιρεία ε, έχει φέρει αυτό το βάρος της απόδειξης ε, και πρέπει να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί δεν είναι σωστοί. Μην τα μπερδεύετε αυτά τα δύο. Δεν μπορείτε να πείτε ότι από εδώ και, το, από εδώ και πέρα είμαι καταγγέλων. Και οτιδήποτε πω ισχύει. Και θα πρέπει η εταιρεία να αποδείξει ότι αυτά που λέω εγώ δεν είναι σωστά. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ε, προβλέπει κάτι τέτοιο το δίκαιο στα κράτη Γι' αυτό μπορείτε να πείτε όμω ότι αν κάποιο είναι καταγγέλων και υπάρχουν κάποιε κυρώσει εναντίον του, αυτοί που λαμβάνουν κυρώσει εναντίον του, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν ότι δεν τον τιμωρούν, δεν παίρνουν αυτές τις κυρώσει εναντίον του επειδή έγινε καταγγέλων, επειδή είναι καταγγέλων. Διάκριση, ε. Επίσης θα έλεγα ότι ο άμεσος κίνδυνο είναι κάτι συχνά αυταπόδεικτο. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να περιμένεις μήνες για να κάνεις κάτι. Λόγω θέματων δημόσια υγείας, λόγω οικονομικών συμφερόντων, όλα αυτά τα οποία παριθμούμε στον κατάλογο ε, μπορεί να πληγούν. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με αυτά. Γιατί η, η βλάβη στα συμφέροντα των φορολογουμένων ή στην υγεία του κοινού κτλ. είναι τόσο μεγάλες, ε, οι ζημιές αυτές τόσο μεγάλες και τόσο προφανείς κτλ. που δεν μπορεί κανείς να περιμένει. Για την προστασία στον χώρο εργασίας που εντάσσεται ε, στους εργασιακούς νόμους. Εκτιμούμε ότι η προστασία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι σε υψηλότερη θέση από την προστασία που προσφέρουμε μέσω της οδηγίας για τους καταγγέλλοντες και την προστασία των καταγγελόντων. Μην τα μπερδεύετε αυτά δύο. Εάν χρειάζεται να αυξήσουμε την προστασία, αν να αυξήσουμε την προστασία ανθρώπων που ε, στο χώρο εργασίας τους, ε, την υγεία και την ασφάλεια. Α το κάνουμε μέσω τη οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια, όχι μέσω τη οδηγία για την προστασία των καταγγελόντων. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσέγγιση, η σωστή. Έπειτα, γιατί χρειάζεται ενωσιακή νομοθεσία. Το παράτημα της οδηγίας απαριθμεί διάφορα θέματα. Αν κάποιος δει ότι υπάρχει μια απειλή στο περιβάλλον, στην ε, ασφάλεια των τροφίμων, στη δημόσια υγεία, στα οικονομικά συμφέροντα κτλ. Ο καθένας το βλέπει αυτό και δεν θα πούν αυτοί αυτή, αν είναι, είναι εθνικό δίκαιο ή είναι ενωσιακό δίκαιο. Όχι. Επειδή επηρεάζει την εσωτερική αγορά, είναι ενωσιακή νομοθεσία. πρέπει να ξέρετε ποια είναι τα γενικά θέματα, ο καθένας πρέπει να ξέρει ποια είναι τα γενικά θέματα που συνδέονται με, την, με τον ενωσιακό δίκαιο. Ας πούμε, δημοσιογεία, η ευμερία των ζώων, οικονομικά συμφέροντα, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, όλα αυτά τα θέματα απαριθμούνται στο παράτημα. Δεν πιστεύω θα υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στην, στο στα επίπεδα δικαίου, εθνικό ή ενωσιακό. Επίσης, ζητάμε τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμίσουν τη δική τους εσωτερική ενωμή τάξη. Αυτή τη στιγμή η πρόταση φτάσει σε επίπεδο διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη, τότε θα μπορούσε η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να κινητοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να ευθυγραμμίσουν την ε, νομοθεσία τους. Γιατί και τα δύο επίπεδα θα εξασφαλίζουν προστασία στους καταγγέλλοντες, ε, αν υπάρξει αυτή η αφιγράμμιση. Αυτά σε, όταν φτάσουμε στις διαπραγματεύσεις. Τώρα, για τις κόκκινες γραμμές. Δεν σκοπεύω να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αρχή. Το θέμα είναι τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό που πρέπει. Εάν δεν το κάνουν, τότε μπορούμε να προσφύγουμε εναντίον τους ε, στο δικαστήριο. Έτσι δουλεύει το ενωσιακό δίκαιο. Και θέλω να σας πω ότι, και με βάση την πρόσφατη εμπειρία, ότι δεν θα διστάσω ούτε μία στιγμή να προσφύγω αντίον ενός κράτους μέλους εάν δεν κάνει αυτά που επιτάσσει η οδηγία. Δεν θα διστάσω ούτε στιγμή. Είναι σημαντικό, γιατί δημιουργείται έτσι ένα προηγούμενο, μια πρακτική ας πούμε, εάν δεν το κάνω. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Λεποετού ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν, θα πρέπει να βελτιώσουν τις πρακτικές, θα πρέπει να δείξουν ότι καταλαβαίνουν ότι η προστασία των καταγγελώνων είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Και υπάρχει και νοσιακή νομοθεσία που ε, εξασφαλίζει ένα πλαίσιο. Και αν δεν εφαρμόσουν οδηγία τα κράτη-μέλη, τότε υπάρχει από πίσω το ενωσιακό δίκαιο που ε, χάρη σε αυτό μπορούμε να προσφύγουμε εναντίον του. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζομαστε και χωριστή αρχή για να το κάνουμε αυτό. Η Κομισιόν μπορεί κάλλιστα να προσφύγει εναντίον ε, ενό κράτου μέλου χωρί να δημιουργηθούν νέοι οργανισμοί. Η νομική βάση που επιλέξαμε, η συγκεκριμένη νομική βάση, το άρθρο 114 μας δίνει τη δυνατότητα να μην καλύπτουμε ανθρώπους μόνο που έχουν σχέση υπαλληλική, που είναι εργαζόμενοι, αλλά να αφορά και ανθρώπους που δεν είναι υπάλληλοι, που είναι μαθητευόμενοι ή που είναι συμβασιούχοι ή που έχουν μια οποιαδήποτε σχέση μη υπαλληλική, μη, που δεν είναι μόνιμη ας πούμε. Και αυτοί θεωρούνται καταγγέλτε. γι' αυτό διάλεξαμε αυτή την νομοθεσία. Το έχουμε τσεκάρει και διπλότσεκάρει μάλιστα το θέμα αυτό. Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε αυτό, με ρωτήσατε, και την, περίπτωση, και την υπόθεση Σελμάιερ. Πώς μπορείτε να τα συνδέσετε αυτά τα δύο. Αλλά ο κ. Λεμπρετό μπορεί να μα εξηγήσει, μπορεί να μα πείσει. και μπορεί να προσφύγουμε στην ε, νομική υπηρεσία του, Κοινοβουλίου, το οποίο ε, έχει διερευνήσει αυτή την υπόθεση. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέση. Πάμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Κύριο Ράντιεφ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμανς, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα για να απαντήσετε ερωτήσεις και παραδοχόμενες και οι προσπάθειες της ε, Κομισιόν τα τελευταία χρόνια. Η Κομισιόν έχει κάνει πολλά βήματα για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα στην νομοθεσία και στην πολιτική. Και είμαι σίγουρος ότι έτσι η νομοθετική διαδικασία θα γίνει πιο προσβάσιμη και θα ενσωματώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών. Ένα από αυτά τα βήματα όταν μιλάμε για την αναθεώρηση της νομοθεσίας ήταν ο σχηματισμός μιας ομάδας εργασίας για την αναλογικότητα, την επικουρικότητα και το πώς θα κάνουμε λιγότερα πράγματα πιο αποτελεσματικά. Στην τελευταία ολομέλεια εγκρίναμε μια έκθεση του Κοινοβουλίου για τις αιτήσιε εκθέσεις για την εφαρμογή των αργών της επικουρικότητας και αναλογικότητα για το 2015 και 2016. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Task Force αυτής. Αναμένω και την έκθεσή σας που θα δημοσιευτεί το καλοκαίρι. Έχει βρει η ομάδα εργασίας κάποιους τομείς που υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επίσης θεωρείται ότι η εισαγωγή περισσότερης ευελιξίας όταν μιλάμε για την ε, περίοδο αυτή των 8 εβδομάδων που έχουν τα κράτη-μέλη για να αντιδράσουν σε νέε νομοθετικέ προτάσει. θα ενισχύσει τον ρόλο του ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Κύριος Σβιεύκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για τις εξηγήσει του και ευχαριστώ και για τις ισορροπημένες αυτές προτάσεις το σκεπτικό είναι να δούμε ακριβώ ποιος είναι καταγγέλων και τι προστασία πρέπει να τύχει. Περνάμε τώρα στα υπόλοιπα. Για το εταιρικό δίκαιο και εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την νομοθεσία που προετοιμάζεται, αλλά βεβαίως ε, έχουμε ένα έτος ακόμα μπροστά μας νομοθετικής εργασίας και η τελευταία μας συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του επόμενου έτους και έχω κάποιες ανησυχίες για το εάν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το νομοθετικό μας έργο και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βεβαίως εμείς θα καταβάλουμε όποια προσπάθεια γίνεται, αλλά θα δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση του Συμβουλίου. Τώρα, περνάω στις ερωτήσεις. Ο κ. Σαέρα μου ζήτησε να κάνω κάποιες ερωτήσεις εκ μέρου του. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν αφορά την δουλειά η οποία γίνεται στο πολιτέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Μια ερώτηση άμεση προς εσάς κύριε Αντιπρόεδρε. Θα θέλαμε να μας διαβεβαιώσετε δημοσίως πως οι αρμοδιότητες ε, του Κοινοβουλίου στις πράξεις κάθε εξουσιοδότηση και κάτι εφαρμογή θα διατηρηθούν για να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε με την δουλειά μας. Και το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελε να θέσει ο αφορά το Omnibus. Τώρα βεβαίω τρέχουμε, αλλά Κοινοβουλίου θα θέλει να πάει πιο γρήγορα παρόλα αυτά στο πολιτικό επίπεδο. Οπότε το ερώτημα το εξή. Η προθεσμία της 3ης ε, Μαΐου είναι μια προθεσμία την οποία θα τηρήσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σντουιρό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμαντ, ήθελα να πάρω το λόγο πρώτα απ' όλα να σα συγχαρώ για το εξαιρετικό έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετέχα κάποια ανησυχία, γιατί σα άκουσα να λέτε ότι συμφωνείτε με τον κύριο Λεμπρετό. Και ξαφνικά ο ενθουσιασμό μου έπεσε. Άρχισα να λέω, μα τι γίνεται. Αν πράγματι η πρώτη αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερίζεται την άποψη του Εθνικού μετόπου, ε, έχω αμφιβολίες ή ξαφνικά και πολύ χαίρομαι αν το εθνικό μέτωπο προσεγγίζει πιο ευρωπαϊκές απόψεις και ελπίζω, φυσικά ελπίζω, Τέλο πάντων. Στην πραγματικότητα για αυτή την υπόθεση θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ. Δεν έχω σχόλια επί της αρχής. Θα ήθελα να βάζαμε στο ίδιο επίπεδο την προστασία των καταγγελόντων με την ε, ε, προστασία του εμπορικού απόρριτου. Να υπάρχει διαφάνεια. Τι ξέρετε τη θέση μου. Δεν μπορέσαμε να έχουμε πλειοψηφία για αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο. Πάντως σας ευχαριστώ για ό,τι κάνατε μέχρι τώρα. Και σας ευχαριστώ ε, που θελήσατε να βάλετε και το θέμα της πρόθεσης Κοιτάξτε, αυτή η προστασία θα κινδύνευε αλλιώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν και μπορείτε να είσαστε βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει το κείμενο αυτό και για να το βελτιώσει. Και ακριβώς για το θέμα της Ευρωπαϊκής Αρχής και ανεξάρτητα από την παρατήρηση που έκανα στην αρχή, την κάπως ανεκδοτική. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να συμπεριλάβει το ευρωπαϊκό δίκαιο στην εθνική νομοθεσία, έτσι. Οπότε να υπάρχει στο εθνικό δίκαιο η προστασία των καταγγελόντων. Όμως έχω ένα πρόβλημα και το είδαμε ότι η νομοθεσία του Λουξεμβούργου, για παράδειγμα, προέβλεπε την προστασία των καταγγελόντων, αλλά όχι την ε, παραβίαση ενός εθνικού κειμένου για να προστατευτούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω εδώ πέρα νομικίστικες ε, παρατηρήσεις, αν και είμαστε στην Νομική Επιτροπή. Πάντως, από τη στιγμή που αυτή η οδηγία θα τεθεί σε εφαρμογή και θα εφαρμοστεί στις διάφορες χώρες ε, μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πάνω από την εθνική νομοθεσία. Και εκείνο που θέλω να διευκρινίσω αυτό που είπε ο κ. Λεμπέτον, δηλαδή, είναι η μόνη περίπτωση όπου οι εθνικέ αρχέ, είτε δικαστικέ είτε ανεξάρτητε, δεν πρέπει να μπλοκάρουν στο όνομα του συμφέροντο του κράτου το δίκαιο τη Ένωση. Και συγγνώμη που επιμένω και θέλω να είμαι ακριβή γι' αυτό, γιατί όντω τι λεπτομέρειε εφαρμογή του κειμένου αυτού θα κρυφούν όλα. Και κάτι τελευταίο. Επιμένω δεν ακόμα, αλλά θα έπρεπε. Ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εκείνο της ΦΑΡΣ. Είναι γνωστό, είναι μια μεγάλη γαλλοελβετική επιχείρηση η οποία χρηματοδότησε για να μπορέσει να συνεχίσει τις δραστηριότητε της σε χώρες σε πόλεμη κατάσταση και χρηματοδότησε την ΤΕΣ για να μπορέσει να δουλέψει εκεί. Το ξέρουμε. Λοιπόν, ειλικρινά δεν βλέπω πώς μπορούμε με μια εσωτερική διαδικασία, εφόσον είναι γνωστά τα γεγονότα, δεν βλέπω ποια εσωτερική διαδικασία, σε ποια επιχείρηση θα είχε τη δυνατότητα και την αρχή να πάει στις διευθυντικές αρχές, είτε πρόκειται στη δικάτη του οποιοδήποτε θέλει και να τους πει, κοιτάξτε, προσέξτε, αυτά που κάνετε δεν είναι καλά, χρηματοδοτείτε κτλ. Γιατί είναι το γενικό συμφέρον της επιχείρησης να συνεχίζει τις δραστηριότητές της και να μπορέσουν έτσι να συνεχίσουν την εργασία τους και οι εργαζόμενοι. Οπότε επιμένω πραγματικά ότι δεν πρέπει να βάζουμε ιεραρχία στι εσωτερικέ διαδικασίε. Δεν λέω να μην υπάρχουν στις μεγάλες επιχειρήσει εσωτερικέ διαδικασίε, να υπάρχουν, αλλά να μην τι ιεραρχούμε. Γιατί είναι πολλά μεγάλα ζητήματα τα οποία θίγουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Και σε αυτέ τι περιπτώσει δεν μπορούμε να περιοριστούμε στι εσωτερικέ διαδικασίε ούτε μπορούμε να καθυστερούμε με τι ε, καταγγελίε στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Όταν τεθεί το θέμα των αποδείξεων, είναι προφανές ότι σε εσωτερικές διαδικασίες, όπως με το Dieselgate, οι αποδείξεις μπορεί να κρύβονται, να καλύπτονται και να εξαφανίζονται. Οπότε στηρίζω την Επιτροπή να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε λιγάκι αυτό το σημείο και να φροντίσουμε η εσωτερική διαδικασία να μην είναι υποχρεωτική για τους καταγγέλλοντες. Και αυτό που είπε και ο Ζούλιαν πριν, για την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Κύριε Τίμερμαντς, και εγώ έχω μια σύντομη ερώτηση. Στην αρχή αναφερθήκατε στη δημοσιογραφία. Συνδέεται τη δημοσιογραφία με το κείμενο αυτό. Για εξηγήστε μου πώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ξέρετε, αν ε, ε, κατεβάσει καμιά καλή ιδέα το εθνικό μέτωπο, πρώτον θα εκπλαγώ. Αλλά δεύτερον πρέπει να πω ότι είναι καλή ιδέα. Αυτή θα είναι η στάση μου. Ε, τώρα, να σοβαρευτούμε. Η Task για την επικουρικότητα που με ρώτησε ο κύριος Ράντεφ. Πρώτα απ' όλα, λυπούμε για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μην ε, λάβει μέρος ε, στην Επιτροπή αυτή γιατί θα ήσασταν πιο ενήμεροι από ό,τι είστε τώρα και βεβαίως ε, θα συνεισφέρατε και στο έργο της Επιτροπής που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό γιατί τα Εθνικά Κοινοβούλια που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται, έχουν πολλά έγγραφα, πολλές ιδέες και η Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι πολύ δραστήρια εκεί. Είναι σε επαφή με τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές και ξεκαθαρίζει το πώς μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερες επαφές ε, στην κοινοτική νομοθεσία και είναι πολύ σημαντικό για μας να ακούμε τους πελάτες μας εντός εισαγωγικών για το πόσο δύσκολο είναι να εργαστούμε αυτή την νομοθεσία και το πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την διαδικασία αυτή και να εντάξουμε αυτές τις ιδέες ε, εξ αρχής ε, στην ομοθέσια Γιατί αυτό το οποίο προξένει σε έκπληξη είναι ότι ο κόσμος ε, έχει πρακτικές ιδέες. Πρέπει να τα εφαρμόσουν αυτά. Μιλάνε στους επιχειρηματίες επιτόπου Πρέπει να φροντίσουν αυτά τα πράγματα να είναι εφικτά για τους ε, πολίτες. Και έτσι θα έχουν ε, βεβαίως ε, αποτελέσματα, γιατί συχνά κατηγορείται η κοινοτική νομοθεσία, χωρίς να φταίει, για το ότι τα πράγματα είναι περίπλοκα. Το να το συζητάμε λοιπόν μαζί τους. Και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις είναι προς το όφελος όλων μας. Οπότε οτιδήποτε και αν γίνει πριν ε, γράψουμε την έκθεση. Αυτή τη στιγμή στην γράψουμε, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα είναι σε επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης. Αυτό νομίζω θα μας ωφελήσει όλους. Και πάλι να τονίσω ότι ο τρόπος ε, με τον οποίο είναι σε επαφή μαζί μας οι εθνικές αρχές, ε, τα κοινοβούλια, δεν αφορά μια συζήτηση για το φύλλο των αγγέλων, για το τι εστί η επικουρικότητα. Έχω βαρεθεί πια αυτές τις συζητήσεις, ε, τις είχα κάνει και με την προηγούμενη ιδιότητά μου, γιατί βεβαίως ο καθένας ε, καταλαβαίνει ότι θέλει με την λέξη αυτή. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άλλες αρχές ε, για να εργαστούν καλύτερα για το τι πρέπει να νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες που έχουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες μας και επίσης σε ποιους τομείς θα πρέπει να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετεί ή να ζητήσει νέα μέσα για νέες προκλήσεις. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει και θα συνεχίσουμε να τα συζητούμε και με τους ειδικού, θα ζητάμε ενημερώσεις. Παραδείγματος χάρη είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά από τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού ήρθε και μας μίλησε για τα όρια του Ευρωπαϊκού Δικαίου που πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Μα κάθε σεβασμό. Κανείς δεν μιλάει για αφαίρεση αρμοδιοτήτων. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια συνεργασία με τρόπο που ελπίζουμε να βρει στήριξη στους πολίτες, τους ανθρώπους για τους οποίους δουλεύουμε τελικά. Αυτά λοιπόν θέλουμε να γίνει κάτι με τρόπο ρεαλιστικό, συγκεκριμένο, με συνεργασία και ελπίζω μέχρι τον Ιούλιο να έχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα γραπτός για το εταιρικό δίκαιο. Να τονίσω ότι, ξέρετε, έγιναν πολλές απόπειρες τα τελευταία 15 χρόνια να βελτιωθεί το εταιρικό δίκαιο και καμία φορά τελικά δεν είχαμε αποτέλεσμα. Ελπίζω αυτή τη φορά να φέρουμε μια πρόταση η οποία θα πετυχαίνει την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας στην εσωτερική αγορά χωρίς η ευελιξία αυτή να είναι εις βάρος των εργαζομένων ή άλλων συμφερόντων που πρέπει να προστατευτούν. Αυτή είναι η ισορροπία που αναζητούμε. Ευελιξία ναι, αλλά όχι εις βάρος του φορολογούμενου και των εργαζομένων που εργάζονται και θα επηρεαστούν εάν η εταιρεία αλλάξει έδρα. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτά τα πράγματα για να πετύχουμε την σωστή λύση. Είναι αυτή η σωστή λύση. Θα δούμε, θα το θέσουμε τόσο θα γίνει μαζί σας μια συζήτηση και θα δούμε πού μπορούμε να πάμε. Για το πι δελτα πι. Με εξέπληξε η ερώτηση για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και κατά εφαρμογή. Θα προτείνουμε γι' αυτό το καταλληλότερο, το μέσο ε, και κατά περίπτωση. Από ό,τι είδα, δεν υπάρχει πρόθεση και θα σας το διορθώσω αν ε, δεν έχω δίκιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε την ε, κατανομή ευθυνών ε, ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα μέσω κατεξιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων. Ε, θα το τσεκάρω, όμως θα το δίπλο τσεκάρω και αν χρειαστεί θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Τώρα, για το θέμα των καταγγελόντων. Αν αυτή η οδηγία ε, υιοθετηθεί υπό την ε, παρούσα της μορφή από όλα τα κράτη-μέλη, τότε η λουξεμβουργέζικη νομοθεσία σε αυτή την περίπτωση δεν θα προσφέρει διέξοδο. Κάποιος ας πούμε ότι που κατήγγειλε ε, φοροδιαφυγή δεν σημαίνει ότι δεν θα προστατεύεται. Αν εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, θα θεωρηθεί αυτό το άτομο ως καταγγέλλον και θα απολαμβάνει τις ε, προστασίες. Και όπως ξέρετε, εδώ πριτανεύει το ενωσιακό δίκαιο και επομένως ισχύει η οδηγία. Δεδομένης της ε, φύσης της ερώτησής σας και δεδομένης της ε, γνώσης που έχετε στον τομέα, χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε για να το διευκρινίσουμε αυτό και να κάνουμε μια συζήτηση επίσης γι' αυτό. Ε, και εγώ θέλω να το επιβεβαιώσω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ούτω ή άλλω στη συζήτηση που θα κάνουμε θα το διευκρινίσουμε 100% για τι εσωτερικέ διαδικασίε. Πάντα αυτό θα είναι δύσκολη επιλογή. Το να έχουμε μια ιεραρχία που να λέμε πρώτα εσωτερικά κανάλια, εν συνεχεία δημόσιε αρχέ, δημόσιοι φορεί και αν δεν πετύχει αυτό που θέλει, δεν, πάρεις, ε, δεν ικανοποιηθεί, μπορεί να προσφύγει ε, στον τύπο και να τα πει όλα αυτά στο κοινό, α πούμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή δομή, αλλά δέχομαι ότι αν ένα καταγγέλλον σκέφτεται ότι αν εγώ πάω, ας πούμε, στις, στα εσωτερικά κανάλια, ε, θα κρύψουν τις αποδείξεις, εάν πιστεύει κάτι τέτοιο ο καταγγέλων και αποφασίσει να πάει στο κοινό, επειδή θεωρεί ότι δεν θα δικαιωθεί με τα εσωτερικά κανάλια και να πάει κατευθείαν δηλαδή στο κοινό, Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η οδηγία προσφέρει την ευελιξία στον καταγγέλλοντα να εξηγήσει με επιχειρήματα και να εξηγήσει ότι αν δεν το είχα κάνει απευθεία αυτό, θα με είχαν εμποδίσει, θα με είχαν θυμώσει ε, και θα είναι πολύ δύσκολο στου άλλου να διασκεδάσουν ε, και να αντικρούσουν αυτό το επιχείρημα. Αλλά σα φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο αποφεύγει ε, τις ελαφρά την καρδία καταγγελίε από οποιονδήποτε α πούμε ε, κάποιο ο οποίο προσφεύγει κατευθείαν στον τύπο και στο χοινό, ε, τη στιγμή που υπάρχουν εσωτερικέ διαδικασίε και δεν τι χρησιμοποιεί παρόλα αυτά. Θα πρέπει, σε περίπτωση που απευθύνεται κατευθείαν στον τύπο, α πούμε, προ τα έξω, να πρέπει να μπορεί να αιτιολογήσει τη στάση του. Τα παραδείγματα που υπάρχουν, συμφωνώ ότι δείχνουν ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ένας καταγγέλων να πει Κοιτάξτε, είμαι πεπισμένο ότι αν προσφύγω στην εσωτερική διαδικασία θα κρύψουν τι αποδείξει ή οι αποδείξει αυτέ θα εξαφανιστούν. Τότε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προσφεύγει απευθεία στο κοινό. Αλλά θα πρέπει να έχει επιχειρήματα για κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να λέει κάνω ό,τι θέλω, οποιαδήποτε από τι τρει οδού. Διαλέγω οποιαδήποτε από τα, οποιοδήποτε από τα τρία κανάλια ας πούμε υπάρχει. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση της διαδικασίας, θα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια πλαισίωση της διαδικασίας. Θα το κοιτάξω όμως ξανά όταν το συζητήσουμε αυτό. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να τελειώσουμε πριν το τέλος των, της εντολής του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και ελπίζω να εγκριθεί. Η τελευταία ερώτηση του Προέδρου για τα συμφέροντα των δημοσιογράφων. Μην ξεχνάτε ότι οι δημοσιογράφοι είναι και αυτοί εργαζόμενοι. Αν πιστεύουν ότι πρέπει να καταγγείλουν κάτι ε, για αυτά που συμβαίνουν στη δική του οργάνωση, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα. Αλλά τέλο πάντων δεν είπατε αυτό. Η, θέση, η ερώτησή σα ήταν ποια είναι η σχέση του με του καταγγέλλοντε. Κοιτάξτε το LuxLeaks. Τα Panama Papers. Το σκάνδαλο με του διτζαλοκινητήρε και το Cambridge Analytica πιο πρόσφατα. Μιλάμε για θαραλέους ανθρώπους που πήγαν και μίλησαν σε δημοσιογράφους. Αν εγώ είμαι δημοσιογράφος και θέλω να συνομιλήσω με κάποιον, και διαρωτώ με, θα πρέπει να το κάνω αυτό, ε, γιατί αυτή η δουλειά έχει και τα ρίσκα της. Αν καταλαβαίνετε ότι αν ξέρω εγώ ότι το άτομο αυτό θα προστατευτεί από το δίκαιο ή από τις αρχές ας πούμε, ε, θα διαφοροποιηθεί, θα, αλλάξει και η στάση των δημοσιογράφων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δημοσιογράφοι κατήγγυλαν μια ιστορία και καταστράφηκαν από το γεγονός ε, που, ότι ο καταγγέλλοντας που τους αποκάλυψε αυτά τα πράγματα απολύθηκε, τιμωρήθηκε ή βρέθηκε σε πάρα πολύ δεινή προσωπική κατάσταση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυτολογοκρισία του δημοσιογράφου. Αν ξέρει όμως ο δημοσιογράφος ότι προστατεύονται καλύτερα τα άτομα αυτά που καταγγέλουν, τότε αισθάνονται πιο ελεύθεροι δημοσιογράφοι να τα δημοσιοποιήσουν όλα αυτά στο κοινό, να γράψουν την ιστορία για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρώτη Αντιπρόεδρε Τίμερμανς που ήρθατε και απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Σωστά μειώσατε το χρόνο της αρχικής σας παρουσίασης γιατί να με τις ερωτήσεις εξαντλήθηκε ο χρόνος. Ελπίζουμε να σας δούμε το αργότερο στην ακρόαση της κυρίας Χαουτάλα, έτσι. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης ΕΑΒΑ με θέμα μια κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους κανόνες χρειαστικής ευθύνης και την ασφάλιση για συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα. Θα μιλήσω λουξεμβουργικά για να φύγετε από την αίθουσα μου φαίνεται. Φαντάζεστε ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που επιτέλους έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης. Λοιπόν, έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης. Πού είναι η Τατιάνα όμως. Α, εκεί στο βάθος θα μας παρουσιάσει τη μελέτη και μπορούμε να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Για να έχουμε και χρόνο για σχόλια. Τατιάνα, έχετε τον λόγο. Thank you and good afternoon. I apologize. Ευχαριστώ. συγγνώμη που δεν μπορώ εγώ να αλλάξω τις διαφάνειες από εδώ. Θα ακούνα το χέρι μου για να αλλάζει. Είναι δύσκολο βέβαια μετά τον Τίμερμανς ε, να παίρνει κανείς το λόγο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τα πράγματα και ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε. Αυτή η εβδομάδα είναι ιδιαίτερη και είναι πολύ επίκαιρη η παρουσίαση της έκθεσης αυτής, πιστεύω, γιατί αυτή τη βδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει στρατηγική όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι λοιπόν πολύ καλό που έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε θέματα που έχουν να κάνουν περί ευθύνης και την ασφάλιση για συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα. Η Επιτροπή σας είχε νωρίτερα ψήφισμα για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Δελβό και είχε υπάρξει και δημόσια διαβούλευση. Οπότε προσέξτε με για ένα λεπτό παρακαλώ για να σας πω ποια είναι τα στοιχεία κλειδί ευρήματα της έκθεσης αυτής. Τη έρευνα αυτή. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση και πολύ γρήγορα μάλιστα για θέματα ευθύνης και η Επιτροπή σας ημερίζεται αυτή την άποψη από όσο ξέρω. Τώρα, στην έρευνα αυτή εξηγούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Πρώτον, ποιο είναι το γενικό πλαίσιο πολιτικής και γιατί χρειάζεται δράση. Μετά βλέπουμε ποια είναι η τρέχουσα ευρωπαϊκή ρύθμιση και εντοπίζουμε τις αδυναμίες, τις ελλείψεις της σημερινής νομοθεσίας. Μετά θα εξηγήσω ποιες θα μπορούσαν να είναι κάποιες προτάσεις για ενωσιακή δράση και τέλος, αντί συμπεράσματος, θα σας παρουσιάσω τις πρώτες εκτιμήσεις για το τι θα μπορούσε να ήταν η Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Εξή εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλάβει δράση. Εδώ βλέπετε πώς καταλήξαμε στην εκτίμηση αυτή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας βασιστήκαμε στο έργο και της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου γενικότερα. Τώρα θέλω να επικεντρωθώ λίγο στην επόμενη διαφάνεια γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει δράση. Τρία ζητήματα τίθεται εδώ. Το πρώτο είναι οι οικονομικές δυνατότητες που θα μπορούν να έχουν η ευρωπαϊκή βιομηχανία και η ευρωπαϊκή κοινωνία γενικότερα. Και εξηγούμε στην έκθεσή μας διάφορα στοιχεία από πού δηλαδή απορρέει αυτή η προστιθέμενη αξία και τα οικονομικά ωφέλη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και είναι και πολύ ανταγωνιστική. Για να καταλάβετε το μέγεθος της βιομηχανίας, η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία απασχολούν 12,6 εκατομμύρια ανθρώπους. 9 φορές δηλαδή περισσότερο από τον πληθυσμό ολόκληρη της Εσθονίας, της δικιάς μου χώρας. Και προβλέπω ότι το 2050 θα έχουμε 17 τρισεκατομμύρια ευρώ ε, με το οποίο θα συνεισφέρει η αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό και θα πρέπει να φροντίσει να υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα που υπάρχει. Τώρα, μιλώντα για αυτέ τι οικονομικέ δυνατότητε, από την ξέρουμε ότι το κοινό ανησυχεί πολύ για το θέμα. Έχουν γίνει διάφορε μελέτε που προσπαθούν να εκτιμήσουν κατά πόσο το κοινό είναι έτοιμο για αυτόνομη οδήγηση. Και μετά από διαβούλευση που κάναμε πέρυσι, φάνηκε ότι 87% των όσων απάντησαν πιστεύουν πως πρέπει να ληφθεί η ρυθμιστική δράση για τα οχήματα αυτά. Ήταν ε, η πρώτη ανησυχία βασικά των πολιτών όταν τους ρωτούσαμε για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Και 74% είπαν ότι τα περιευθύνης είναι μία από τις κυρίες ανησυχίες τους. Συνεπώς, πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο θα έπρεπε να αναλυφθεί δράση. Και το τρίτο που θέλω να σας πω σχετικά με το γιατί πρέπει να αναλυθεί η δράση, αυτό απορρέει από την ανάλυση των ε, αδυναμιών και των κενών που υπάρχουν στην τρέχουσα νομοθεσία. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο περί Ξεκίνησα πριν λέγοντάς σας ότι επιγόντως χρειάζεται δράση, εδώ και τώρα. Αυτό βασίζεται σε δύο πράγματα πρώτα απ' όλα στις ποιοτικέ αλλαγές. Η αυτόνομη οδήγηση δεν θα είναι η ενίσχυση ενός προϊόντος που ήδη υπάρχει, η επέκτασή του. Όχι. Θα πρόκειται για κάτι εντελώ καινούριο. Θα μοιάζει με κοινό αυτοκίνητο, αλλά δεν θα είναι. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Είναι λιγάκι όπως όταν περάσαμε από το άλογο στο αυτοκίνητο. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη διαφορά σημαίνει αυτό. Τώρα, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στα περιευθύνης. Σήμερα βασιζόμαστε για το κίνδυνο σε δύο υποθέσεις. Πρώτον, ότι μπορεί να χαλάσει κάτι στο hardware, στο, στα δομικά υλικά, τέλο πάντων, του οχήματος, και αυτό καλύπτεται από την οδηγία για την κάλυψη προϊόντος. Και το δεύτερο είδος κινδύνου έχει να κάνει με τη δράση του οδηγού. Και εδώ εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες, οι οδικοί. Το όχημα όμως χωρίς οδηγό γίνεται σαν έναν υπολογιστή παντοδύναμο που μας βοηθάει να πάμε από το σημείο α στο σημείο β. Οπότε, αν υπάρξει κάποια δυναμία, δεν έχει να κάνει μόνο με τα δομικά υλικά, έχει να κάνει με το λογισμικό, έχει να κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ πιο περίπλοκα, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια δυναμία κατά την οδήγηση. Το άτομο που βρίσκεται στο αυτόνομο όχημα μπορεί να ονομαστεί οδηγός παραδοσιακά, οπότε να ισχύουν και οι κανόνες οι εθνικοί, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι ισχύει όσον αφορά την ασφάλιση του οχήματο. Τώρα πολύ σχηματικά εδώ λέω ποιε είναι οι αδυναμίες και τα κενά της νομοθεσίας. Στην έκθεση θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτά. Εδώ θα αναφερθώ μόνο σε μερικά στοιχεία. Γενικά μιλώντας έχουμε δύο ζητήματα εδώ. Το ένα έχει να κάνει με τα σημερινά κενά της νομοθεσίας που σημαίνει ότι χρειάζεται να αναλυθούν. Και το δεύτερο είναι νέοι κίνδυνοι που υπάρχουν και που δεν καλύπτονται καθόλου από την τρέχουσα νομοθεσία. Και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά. Τώρα γιατί πιστεύουμε ότι η οδηγία για την κάλυψη προϊόντος δεν φτάνει. Η οδηγία για την κάλυψη προϊόντος είναι μια νομική πράξη που χρειάστηκε μάλιστα χρόνια να συμπεριληφθεί στην νομοθεσία. Και οι ενδιαφερόμενοι πιστεύουν ότι προσφέρει κάποια προστασία, κάποια ισορροπία απέναντι στους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Όμως όσο πιο περίπλοκο γίνεται το προϊόν, τόσο λιγότερο ανταποκρίνεται η οδηγία αυτής της ανάγκης. Ένας περιορισμός από την οδηγία αυτή για την κάλυψη προϊόντος είναι ακριβώς γιατί πρόκειται για μια γενική οδηγία που καλύπτει πράγματα από πολύ απλά ένα μολύβι μέχρι ένα πολύ περίπλοκο προϊόν. Και η βασική ιδέα της οδηγίας αυτής για την κάλυψη προϊόντος είναι όταν υπάρχει κάποιο λάτωμα στο προϊόν. Μόνο λατωματικά προϊόντα τη στιγμή που βγαίνει το προϊόν από το εργοστάσιο ε, μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοια ασφαλιστική κάλυψη. Για να το αποδείξει όμως ο καταναλωτής αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελωτηματικό τη στιγμή που το όχημα βγήκε από τον ημάντα παραγωγής. Και επειδή το αυτόνομο όχημα είναι ένα πολύ περίπλοκο προϊόν που έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα, με την παραγωγή, με τον αυτοματισμό κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τα δικαστήρια που θα κληθούν να αποφασίσουν να πούνε ποιο στοιχείο έχει να κάνει με κάτι ελαττωματικό και τι όχι. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Ένα στοιχείο είναι εκείνο που θα επέτρεπε να μπορούν να μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στους παραγωγούς και στην περίπτωση της αυτόνομης οδήγησης. Εμείς πιστεύουμε ότι εφόσον αφαιθούν στην κυκλοφορία τέτοια οχήματα αυτόνομης οδήγησης, αυτά τα ζητήματα θα προκύψουν όλο και πιο συχνά. Τώρα υπάρχει δεύτερη κολόνα εδώ που περιλαμβάνει κινδύνους που ακόμα δεν καλύπτονται, ή μερικώς ή καθόλου. Αν ας πούμε κάτι δεν πάει καλά με το software, με τον προγραμματισμό, Εντάξει, αν δεν φταίει δηλαδή το δομικό στατικό, αλλά φταίει το προγραμματισμός και υπάρξει ένα τύχημα. Ή αν το ατύχημα οφείλεται σε ένα πρόβλημα του δικτύου ή αν οφείλεται σε ένα πρόβλημα προγραμματισμού εξωτερικό. Δηλαδή το πρόγραμμα πρέπει να κάνει μια επιλογή πώς θα αντιδράσει το αυτοκίνητο στη μία στην άλλη περίπτωση. Και βέβαια έχουμε και τον κίνδυνο από το hacking, έτσι, το έγκλημα, δηλαδή στον κυβερνοχώρο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν καλύπτονται απόλυτα. Σε ένα βαθμό ναι με τα δεδομένα, αλλά πολύ περιορισμένα. Ένας δικαστής ή ένας καταναλωτής που θα κληθεί να λύσει τέτοια ζητήματα θα βρεθεί μπροστά σε πολλές αβεβαιότητες, γιατί τα κενά είναι πολλά και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό που βλέπετε δεξιά, δεξιά σε θέματα που έχουν να κάνουν δηλαδή με ε, μειονεκτική θέση στην οποία θα βρεθεί ο καταναλωτής τελικά και θα υπάρξουν πολλές γκρίζες ζώνες. Θα δημιουργηθούν πολλές αβεβαιότητες και θα ερμηνευθούν διαφορετικά οι κανόνες σε διαφορετικές νομολογίες. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε περισσότερες επίμαχες καταστάσεις και περισσότερες ε, δικαστικές διενέξεις κλπ. Τώρα, να δούμε τι γίνεται από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να δούμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση πριν την στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα λέγαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δούμε τουλάχιστον το ψήφισμα το περσινό, ζητάει περισσότερη δράση. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο επιφυλακτική και λέει ας περιμένουμε να δούμε. Ας κυκλοφορήσουν τα οχήματα αυτά και θα δούμε. Μια τέτοια στάση, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν επικίνδυνη. Διότι τα γεγονότα δείχνουν ότι πολύ πιο γρήγορα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά αυτά τα αυτονομοχήματα. Οπότε ανάλογα με το πόσο χρόνο θα πάρει η νομοθεσία μπορεί να είμαστε έτοιμοι πολύ αργά. Άρα θα χάσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και οι χώρες μέλη θα χάσουν αυτήν την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Και τώρα έρχομαι στο επόμενο. Πριν περάσω αυτή καθ' την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, θέλω να συνοψίσω κάποια πράγματα που είπα και πριν. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλάβει δράση, θα πρέπει να κοιτάξει τα εξή. Πρώτον, πώς θα αντιμετωπίσει τις σημερινές ελλείψεις και τα κενά, πώς θα αντιμετωπίσει τους νέους κινδύνους και τι κανόνες διαδικαστικούς χρειάζεται προκειμένου να υπάρξει και να καθοριστεί η ευθύνη μέσα ε, στο νέο πλαίσιο αυτόνομης οδήγησης. Αν λάβουμε υπόψη μας τα κενά της σημερινή νομοθεσίας και τους νέους κινδύνους, αυτή την αξιολόγηση που κάναμε προσπαθήσαμε να εξετάσουμε διαφορετικές πολιτικές επιλογές. Υπάρχουν διάφορες εδώ πέρα ιδεώδεις. Ε, στην πραγματική ζωή μπορεί να υπάρξει συνδυασμός μεταξύ τους σε διαφορετικό ποσοστό. Λοιπόν, μια λύση θα ήταν να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, status quo. Η δεύτερη θα ήταν να αναθεωρηθεί η οδηγία για την κάλυψη προϊόντος έτσι ώστε να καλύψει και πιο περίπλοκα προϊόντα όπως είναι τα αυτόνομα οχήματα και να επιβάλλει την ευθύνη στον παραγωγό. Ε, μια άλλη περίπτωση θα ήταν η αναθεώρηση των εθνικών κανόνων ασφάλισης οχήματος. Και το τέταρτο θα ήταν νέοι κανόνες και υποχρεωτική ασφάλιση. Συνεπώς, έχοντας υπόψη τα κενά στα οποία αναφέρθηκα και τις πολιτικές επιλογές, προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε ποια θα ήταν η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην κάθε περίπτωση πολιτικής. Και εκτιμούμε και ποσοτικά, κάναμε δηλαδή μια ανάλυση κόστους-οφέλους, άπαξ και κυκλοφορήσουν τα αυτόνομα οχήματα. Μόνο το οικονομικό σκέλος, έτσι ποια θα ήταν τα οικονομικά ωφέλη εφόσον έχουμε νομοθεσία η οποία θα διευκολύνει την κυκλοφορία των αυτόνομων οχημάτων πιο γρήγορα στην αγορά. Και βασιζόμαστε και σε ποιοτικά κριτήρια. Πώς δηλαδή να εκτιμήσουμε αυτήν την προστιθέμενη αξία ποιοτικά, όχι ποσοτικά. Και εδώ αναπτύξαμε 7 κριτήρια γι' αυτό. Και τα βλέπετε στη διαφάνεια. Είναι το βάρος ε, της ε, διένεξης επίλυσης διαφορών, η νομική βεβαιότητα κτλ. Υπάρχουν ε, όλα αυτά τα κριτήρια και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τα αποτελέσματα για την προσθεθέμενη αυτή αξία. Να συγκριτικά με τις τέσσερις περιπτώσεις, τέσσερις λύσεις. Βέβαια δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, είμαστε στην αρχή μόνο, κάνουμε μια εκτίμηση για την επίπτωση που θα είχε η κυκλοφορία των αυτόνομων οχημάτων. Και βλέπετε εδώ τις τέσσερις λύσεις, η τέταρτη φαίνεται να είναι προστιμότερη, οι 2 και 3 θα βελτίωναν κάπως την κατάσταση, αλλά όχι αρχικά. Και πάμε στην προηγούμενη διαφάνεια μια στιγμή. Εδώ βλέπουμε την ε, περίληψη λίγο πολύ. Δηλαδή οικονομικά, ποσοτικά, μπορούμε να μιλήσουμε για 148 δισεκατομμύρια ευρώ ωφέλη που απορρέουν από δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα προσέφερε περισσότερη βεβαιότητα για τον παραγωγό, περισσότερη εμπιστοσύνη του καταναλωτή στις νέες τεχνολογίες κτλ αλλά υπάρχουν ε, και τα μη ποσοτικά ωφέλη, το οποίο τα βλέπετε στη δεξιά στήλη. Για να ολοκληρώσω και αυτή την τελευταία μου διαφάνεια, εδώ προσπάθησα να τα συγκεντρώσω όλα ποσοτικά, πώς θα μειωθεί το κόστος, ποια είναι το ωφέλη. Τα βλέπετε εδώ, συγγνώμη που είναι σε μικρά γράμματα. Με δύο λόγια θα έλεγα, ναι, 148 εκατομμύρια, Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι τα μη ποσοτικά ωφέλη, τα οποία οδηγούν σε καλύτερη προστασία του καταναλωτή, σε αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις νέες τεχνολογίες, βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των χωρών μελών, σε δοκιμές, ε, άδειες, ε, λειτουργία αυτών οχημάτων, οπότε δεν θα υπάρχει τόσο κατακαιρματισμός και άρα λιγότερες διαφορές και το κόστος συναλλαγών επίσης θα μειώνονταν. Και τελευταία μου πρόταση είναι ότι εάν δεν αναλυφθεί δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλη αυτή η δυνατότητα προσθέμενης αξίας θα χαθεί και αντίθετα θα δημιουργηθεί περισσότερο κόστο, γιατί αργότερα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό. Ήδη τώρα βλέπουμε ότι οι χώρες μέλη αναλαμβάνουν δράση και όχι μόνο οι Ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο ισχύει αυτό γιατί πολλέ χώρε, ε, οι ομάδες χωρών αναλαμβάνουν δράση οπότε θα χάσουμε το πλεονέκτημά μα αν δεν προχωρήσουμε γρήγορα. Την ολόκληρη μελέτη μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα που σας παρουσιάζουμε εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες που βοήθησαν στην εκπόνηση της μελέτης αυτής, που βασίζεται σε τρεις μελέτες. Μία οικονομική ανάλυση που έγινε από τη Randa Europe και μία νομική ανάλυση που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω, να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το τόσο περίπλοκο αλλά και τόσο ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Τατιάνα για την παρουσίαση. Καλό είναι που ανέφερε ότι βασιστήκατε σε τρεις μελέτε για να ετοιμάσετε τη δική σας. Μία για την νομική ανάλυση, μία για την ε, οικονομική ανάλυση και άλλη μία. Γιατί το ερώτημα, το ερώτημα που θέτουμε είναι ποια, θα είναι ποια είναι η προτιμότερη πολιτική. Ίσως δεν ξέρουμε την απάντηση ακόμα. Καταρχάς, να ρωτήσω τους συναδέλφους αν έχουν ερωτήσεις ή σχόλια στη μελέτη. Αλλιώς να συνεχίσω εγώ. Είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για αυτή τη uh, μελέτη και δεν είμαι σίγουρη αν οι ισχύοντες κανόνες είναι αρκετά καλή για την ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων. Το ΟΣΑ λέει ότι υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο συντονισμού ανάμεσα στις διάφορες δικαιοδοσίες. Ακόμα και για τον έλεγχο των αυτοκινήτων ε, υπάρχουν συγκρουόμενοι κανόνες. Το θέμα είναι βέβαια αν θέλουμε αυτόνομα οχήματα στους δρόμους μας ή όχι. Αν τα θέλουμε όμως, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο το έργο μας. Γιατί αν αλλάξουμε τους κανόνες για την ευθύνη των προϊόντων, δεν θα, θα την αλλάξουμε μόνο, αλλάξουμε το πλαίσιο μόνο για τα αυτοκίνητα, παρότι είναι εξειδικευμένο τομέα, ε, πρέπει να αλλάξουμε, θα αλλάξουμε γενικά το πλαίσιο. Το να έχουμε νέου κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια αισιόδοξη ίσω ε, στάση. Ίσως υπάρχει και πιο εύκολη λύση. Ε, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου, γιατί από ό,τι κατάλαβα, η οδηγία για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, αλλά και οι κανόνες για την ευθύνη στο, στο δρόμο δεν προβλέπουν προβλέπουν μόνο την ευθύνη του οδηγού. Με τα οχήματα τι θα έχουμε οδηγό ούτως ή άλλως. Και αν δεν έχουμε δεν ξέρω ποιος θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ε, δίνει την οδηγία, με δίνει την εντολή στο όχημα, να πάει το σημείο Α στο σημείο Β. Ε, αυτός ε, είναι υπεύθυνο για την πιθανή ζημιά. Δεύτερον, πώς μπορούμε να αποδείξουμε το ελάττωμα σε μια τεχνολογία που εξελίσσεται τόσο πολύ. Συνδεόμενο ερώτημα είναι ποιος είναι ε, ο υπεύθυνος για την αναβάθμιση. Όλοι σας έχετε smartphones και πολύ ε, σύντομα ε, λαμβάνω μηνύματα πολύ συχνά μάλλον λαμβάνω μηνύματα ότι θα πρέπει να αναβαθμίσω το τηλέφωνό μου. Καμία φορά το κάνω και το ξεχνάω. Δεν είναι πρόβλημα στο βαθμό που είναι θέμα λειτουργίας της υπηρεσίας μόνο και το πόσο καλά με εξυπηρετεί. Το θέμα είναι ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ένα εργαλείο, με ένα όχημα, το οποίο ας πούμε μπορεί να προκαλέσει ζημιές, ποιος είναι υπεύθυνο, ο οδηγός, ο οδηγός είναι το σημείο κλειδί, το πρόσωπο κλειδί. Ε, ποιος έχει την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση ζημιάς. Ξέρω ποια, ποια είναι η απάντηση. Σε περίπτωση που έχουμε κατάρρευση του δικτύου. Αν γίνει ατύχημα με το αυτόνομο όχημά μου, και είμαι εγώ ο φυγόμενος ας πούμε. Μπορώ να προσφύγω εναντίον του υπεύθυνου του δικτύου και πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι το δίκτυο και όχι ας πούμε το λογισμικό που φταίει για, αυτό το, για αυτή τη ζημιά. Σταματάω και ελπίζω να μου δοθούν κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που είναι βασικά στην καρδιά της όλης συζήτησης. Με βάση αυτές τις τρεις μελέτες καταλήξαμε ότι η μεταρρύθμιση είναι η καλύτερη ε, λύση. Γιατί όταν αρχίσεις να κάνεις μικρές επιδιορθώσεις ας πούμε, στην νομοθεσία, το πράγμα δυσκολεύει, γιατί είναι αλλοσυνδεόμενα αυτά τα πράγματα. Επίσης, κάτι άλλο, όπως υπόθηκε, ε, σε πολλές δικαιοδοσίες ο οδηγός δεν προστατεύεται. Ε, και ο χειριστής δεν θα προστατεύεται. Και γι' αυτό αλλάζουμε την ε, οδηγία για την ευθύνη. Έχουμε το χειριστή του αυτόνομου οχήματος, ο οποίος είναι κάποιο άτομο, είναι στην κυκλοφορία γι' αυτό. Θεωρούμε ε, ότι ο οδηγός με τη δράση του πάντα παραδοσιακά οδηγεί, ε, δημιουργεί τον κίνδυνο. Εδώ όμως αλλάζει τελείως αυτό το πράγμα. Σε ορισμένα κράτη-μέλη στην έκθεση αναφέρεται μία ανάλυση ε, της κατάστασης διαφόρων δικαιοδοσιών και ε, μια με βάση τον κίνδυνο, μια με βάση το, της, την, το κενό, ας πούμε, την έλλειψη. Ε, ορισμένες δικαιοδοσίες ε, προστατεύουν περισσότερο τον οδηγό, κάποιες α, δικαιοδοσίες δεν προστατεύουν καθόλου, δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση. Ε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα ε, με βάση την οσιακή νομοθεσία ακόμα. Ε, τα κράτη-μέλη δίνουν τις απαντήσεις. Επίσης, η οδηγία για την ε, ευθύνη των προϊόντων τι λέει, ότι όταν έχουμε περίπλοκα προϊόντα είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε την ευθύνη. Ε, επομένως, ε, για τον καταναλωτή είναι πολύ αδυναμή η θέση του ε, σε περίπτωση διαφοράς. Έχουμε το άρθρο 7 με τις διάφορες εξαιρέσεις για την ε, υπεράσπιση του καταναλωτή. Το πρόβλημα λοιπόν υπάρχει, ε, πρέπει να αναλυθεί δράση για να λυθεί στην έκθεση. Καταλήγουμε με βάση νομική ανάτηση, ότι το να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσω της οδηγίας για την ευθύνη των προϊόντων θα είναι δύσκολο και η ε, τροπολογία των εθνικών κανόνων για την ε, ευθύνη σε περίπτωση τροχαίου ε, επίσης θα είναι δύσκολο. Ε, επίσης, δύσκολο θα είναι ε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι υπεύθυνο για την αναβάθμιση. Δύσκολο ερώτημα, το συζητήσαμε ε, υπό τους νέους κινδύνους. Είναι θεά ζώνη. Εξαρτάται από την ερμηνεία του δικαστηρίου. Θα δημιουργήσει πολλές διαφορές πολλέ προσφυγέ στο δικαστήριο, παραδείγματο χάρη, μπορεί να θεωρηθεί αμέλεια. Αν, α πούμε, σου έχουν πει 10 φορέ να αναβαθμίσει και δεν το έχει κάνει, θεωρηθεί, μπορεί να θεωρηθεί αμέλεια. Αλλά και ο παραγωγό θα πρέπει να, δώσει κάποιες, ε, να σου στείλει κάποιε κοινοποίησει, κάποιε γνωστοποίησει, ώστε να το υπενθυμίζει συχνά το σύστημα ότι πρέπει να το κάνει. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, θα πρέπει να ε, ενημερώνουμε τον καταναλωτή ότι είναι υποχρέωση. Και αν δεν το κάνει, α πούμε, έχει ευθύνη και επομένω υπάρχουν συνέπειε. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα για την ε, αναβάθμιση του λογισμικού. Ε, είναι προβληματικό ε, θέμα. Το λογισμικό είναι προϊόν, λένε ορισμένοι. Ε, και είναι, άρα ισχύει η οδηγία για την ευθύνη των προϊόντων. Εάν θεωρήσουμε ότι το λογισμικό είναι προϊόν, με βάση την οδηγία αυτή για την ευθύνη των προϊόντων, τότε μπαίνει το εξή ερώτημα. Ποιο είναι υπεύθυνο, ο παραγωγό του λογισμικού ή ο παραγωγό του αυτονομού σε περίπτωση που υπάρξει προσφυγή, ας πούμε. Και αν ο παραγωγός, ας πούμε, του λογισμικού δεν προβλέψει, ας πούμε, την κατάλληλη χρονική στιγμή αναβάθμιση, τότε προφανώς έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Όλα αυτά τα πράγματα είναι περίπλοκα, γι' αυτό λέω ότι αν δεν επιληθούν, θα δημιουργηθούν πολλές διαφορές στα δικαστήρια και πολλές αβεβαιότητες. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τις ε, γραπτές δηλώσεις ε, είναι η εξή, ότι η ισχύουσα νομοθεσία θα μπορούσε να ρυθμίσει τις διαφορές. Α, σύμφωνοι, αλλά με ποιο κόστος. Κατάρρευση δικτύου. Το θέμα της ε, διασυνδεσιμότητας θα είναι τμήμα του πακέτου που παράγει ο παραγωγός. Ε, αν η, η συνδεσιμότητα είναι τμήμα του προϊόντος, τότε μπορείς να προσφύγεις εναντίον του παραγωγού και να πει ότι έχει ευθύνη. Αν ο παραγωγό όμω πει ότι αυτό είναι ευθύνη ενός τρίτου, τότε φυσικά η οδηγία ε, για την ευθύνη των προϊόντων δεν ισχύει. Υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούμε να επιλύσουμε. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε, θα χρειαστούμε νέα νομολογία σε εθνικό επίπεδο και σε νοσιακό επίπεδο. Και επίση, ε, αν υπάρξουν προσφυγέ στα δικαστήρια, επειδή είναι διαφορετικέ οι δικαιοδοσίε και διαφορετικά τα συστήματα, θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Πολύ ωραία. Σαφέ το συμπέρασμα. Δεν ξέρω αν το συμμερίζονται όλοι. Τουλάχιστον δική σα θέση είναι σαφή. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν. Εάν όχι, σα ευχαριστώ. για την παρουσίαση και ούτως ή άλλως έχουμε και τα έγγραφα οπότε μπορούμε να τα μελετήσουμε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους ε, ειδικού και ολοκληρώθηκε η απολυσματινή μας συνεδρίαση και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Το επόμενο θέμα είναι η συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ.